ότι η Ιταλική δικαιοσύνη θα σεβαστεί απολύτως τι υψηλέ προδιαγραφές που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε περίπτωση εκδόσεως. Ευχαριστώ για το θέμα της εκδόσεως του Τσέζαρη Μπατίστη η συζήτηση έληξε. Έχω έξι προτάσεις ψηφισμάτων που θα ψηφιστούν μετά την ολοκλήρωση της ε, τρίτης και τελευταίας συζητήσεως που είναι γύρω από το Ιράν και ιδιαίτερα η περίπτωση της Νασρίν Σότουντεχ. Έξι συντάκτες. Πρώτος ο κ. Μπέλντερ, 1,5 λεπτό. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Precies een... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από μια εβδομάδα η Σιρίν Εμπαδί έγραφε ένα άρθρο στο New York Times για την Νασρίν Σοτουντέ τη φίλη της που καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλακή και ζητήθηκε να προστατευθεί αυτή η προασπίστια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην, στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν μπορούμε εμείς να ξεχνάμε την κυρία Σοτουντέ και όσους διώκονται στο Ιράν. Έχω μια αναφορά του Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα και ζητώ να ψηφίστε ομόφωνα για την ε, δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης του Ιρανικού λαού. Κυρία Σάκη, για δύο λεπτά. Κυρία Σάκη, ευχαριστώ αναγκαζόμαστε ξανά να μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν μετά την καταδίκη 11 χρόνια φυλάκισης τη ε, ε, Νασρίν Σότουντέ. Της απαγορεύεται επίση η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Δεν υπάρχει πλέον κράτος δικαίου στο Ιράν και είναι πολιτικοποιημένη απολύτω η δικαιοσύνη. Η προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων θεωρείται τώρα ότι στρέφεται κατά του Ιρανικού κράτους η Νασίν Σοτουντέ, δικηγόρο και μητέρα δύο παιδιών, θεωρήθηκε ότι έδρασε κατά της κρατικής ασφαλείας επειδή υπερασπίστηκε μία Ιρανο-Ολλανδή ε, πολίτη η οποία είχε συνομιλήσει με ε, Ολλανδούς ε, διπλωματικούς. Βλέπουμε μπροστά μας ένα ανίσχυρο καθεστώς το οποίο καταπιέζει τους πολίτες ε, της χώρας του αντί να τους προσφέρει δυνατότητες ε, ανάπτυξης. Η κυρία Άστον θα μεταβεί στο Ιράν για να ε, συζητήσει σχετικά θέματα. Οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται έχουν τον ίδιο στόχο. Εγώ ωστόσο αμφιβάλλω ότι θα προσφέρουν οποιοδήποτε επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα θίξουν μόνο τον Ιρανικό λαό, ο οποίος με τον τρόπο αυτό γίνεται όλο και πιο εξαρτημένο από του κληροπυρηνικού τη κυβέρνηση αυτή. Και ενώ έχω τι επιφυλάξει μου σχετικά με τι οικονομικέ κυρώσει, είμαι πεπισμένη ωστόσο ότι κυρώσει κατά ατόμων που είναι υπεύθυνα για την παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων, είτε με ε, την επιβολή θανατικών κυρώσεων είτε βασανιστήριων, θα βοηθούσαν οι κυρώσει αυτέ να σταματήσει η πορεία αυτή και να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ασφαλώ και είναι η αχίλια πτέρνα του Ιρανικού καθεστώτος. Σας ευχαριστώ. Και μιας και έχω το λόγο κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να ζητήσετε από τους τελούς συναδέλφους να είναι πιο σιωπηλοί, γιατί τώρα που τελείωσε το θέμα τους συνδιαλέγονται στην Ολομέλεια στα λεγόμενα πειραδάκια. Ο Πρόεδρος, ακούσατε την ε, κυρία Σάκη, ε, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να είστε ε, να σεβαστείτε την ε, ησυχία της Ολομέλειας. Ο κύριος λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόθεσή μου σήμερα ήταν να συγκρίνω την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με την ναζιστική Γερμανία. Πρέπει να πω όμως ότι πιστεύω ότι κατά πολλού τρόπους τα πράγματα ίσως είναι χειρότερα στο Ιράν. Πάντως έχουν κρεμάσει, έχουν καταδικάσει απαγχωνισμό 65 ανθρώπους μόνο φέτος. 10 απαγχωνίστηκαν χθες. Ε, πρώτα κατασχέθηκαν τα υπερχοντά τους και μετά τους ε, μαστίγωσαν προτού τους οδηγήσουν στην ε, κοιλωτίνα. Ε, έχουν τις περασμένες τέσσερις εβδομάδες απαγχωνιστεί οκτώ τουλάχιστον άτομα. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση για όλα αυτά χωρίς καθυστερήσεις. Έχουμε ακούσει τις απειλές για πυρηνικά όπλα, έχουμε ακούσει ότι η ελευθερία των πολιτών του Ιράν με απειλές, απαρχονισμούς, μαστιγώσεις, ε, ε, κατα... θανατικές καταδίκες, ε, φυλακίσεις παιδιών, βασανιστήρια, συνεχώς η ελευθερία των πολιτών λοιπόν υποβαθμίζεται. Ήδη δύο καταδικάστηκαν σε ακροτεριασμό αυτή την εβδομάδα και την, ερχόμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα και το ίδιο θα γίνει την επόμενη. Η περίπτωση λοιπόν της ε, είναι η περίπτωση μια δικηγόρου που προσπάθησε να σώσει πολλού αθώου που αυτό το φασιστικό καθεστώ είχε καταδικάσει σε θάνατο. Μιλάμε για την παράλογη ποινή τη επταετού κάθριξη σε φυλακή. Ε, οι πραγματικοί εγκληματίε όμως και τύρανοι του Ιράν είναι αυτοί που έχουν αναλάβει την πολιτική εξουσία. Αυτοί πρέπει να απαγωνιστούν και νομίζουν ότι όλοι όσοι του επικρίνουν στη Δύση έχουν κάνει μια διεθνή συνωμοσία εναντίον του για να ανατρέψουν το καθεστώ του. Όχι. Ε, δεν θα πρέπει να αφήσουμε αυτέ τι ε, κακέ, τι δυνάμει του κακού να θριαμβεύσουν, αλλά να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τη δημοκρατία στο Ιράν, προκειμένου να εξηγιάνουμε και τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Ο κύριο Κροτσέτα, λεπτό. Grazie Presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μέσα από το αίτημα για την απολευθέρωση της Ναρίν Σουτουντεχ να παλέψουν για το γκρέμισμα του πιο σκληρού και ματηρού καθεστώτος της ιστορίας. Δεν είναι μόνο μία απειλή για την παγκόσμια ειρήνη, το Ιράν με την απειλή δηλαδή ενός ατομικού πολέμου αλλά και μέσα από μαζικές συλλήψεις, δολοφονίες, βιασμό και βία εναντίον όλων όσων αντιστέκονται στο καθεστώς, δίκες, δίκες φάρσα διακρίσεις ε, κατά των γυναικών και των ομοφιλοφίλων, έλλειψη ελευθερίας έκφρασης και συνεταιρίζεσθε στο στρατόπεδο της ΑΣΡΑΦΤ οι Ιρανοί κρατούμενοι υπόκεινται σε άπειρα βασανιστήρια μέχρι και ακροτηριασμούς στρεβλώνονται οι δικαστικές αποδείξεις, οι μαρτυρίες αποσπώνται με βασανιστήρια και αυτές οι κριτικές δεν στρέφονται κατά του Ισλάμ αλλά κατά του καθεστώτος του Ιράν. Η καταδίκη της Νασρίν Σοντούτε δείχνει για μια ακόμη φορά δικαστική μοχθηρία όπου καταδικάζεται ένας υπερασπιστής των πολιτών και δεν δίνεται στους Ιρανούς πολίτες η ευκαιρία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν αρχίζαμε να κοιτάζουμε το φάκελο των πυρηνικών του Ιράν, θα προσέχαμε ότι η πόρτα έχει κλείσει τελείω ό,τι αφορά τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Η περίπτωση τη Νασρίν Σοδουτέ δείχνει, είναι μια κατάφορη απόδειξη. Ε, τιμωρήθηκε γιατί εργάστηκε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μια πολύ σκληρή ποινή. 11 χρόνια κάθεξη, 20 χρόνια απαγόρευση να ασκήσει το επάγγελμά τη ω δικηγόρο, απαγόρευση να βγει από τη χώρα. Και εδώ δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη περίπτωση. Μιλάμε για μια καλώ σχεδιασμένη στρατηγική από την πλευρά του καθεστώτο τη επίσημη κυβέρνηση του Ιράν, προκειμένου να θυμώσει όλου του αντιρρησίε ε, κατά του καθεστώτο. Ε, οι δικηγόροι, ιδίω οι δικηγόροι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, γνωρίζουν τεράστιε πιέσει. Θα πρέπει να του δείξουμε αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη σε όλου αυτού του τολμηρού πολίτε που δρούν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά τι απειλέ κάθριξη και τα βασανιστήρια. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Ρωμέβα ή Ρουέντα για δύο λεπτά. Λυπούμε πολύ για το γεγονός ότι καλούμαστε πάλι να μιλήσουμε για το Ιράν. Αλλά οφείλουμε, διότι η κατάσταση στο Ιράν είναι απολύτως δραματική. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να επαναλάβει ξανά την έκκλησή του για την απόλυση όλων των ε, πολιτικών κρατουμένων για τα φρονήματά τους που έχουν διαμαρτυρηθεί ειρηνικά μέχρι τώρα. Το Κοινοβούλιο οφείλει να ζητήσει και πάλι από τις Ιρανικές αρχές να σεβαστούν τα παγκοσμίω ε, σεβαστά ανθρώπινα δικαιώματα και να καταδικάσει το Κοινοβούλιο την βαριά καταδίκη της ε, Νασρίν Σότουντε. Για το λόγο αυτό επίσης πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεωρήσει την κυρία καλώς και, καθώς και τους συγκρατουμένους της ως κρατουμένους συνειδήσεως. Πρέπει να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για τις όλες και, όλο και περισσότερες καταδίκες που τελικά οφείλει ε, κανείς να σκεφτεί ότι η παραμονή στο Ιράν σημαίνει τιμωρία για αυτούς που μένουν. Όσοι μπορούν φεύγουν. Πρέπει να ζητηθεί ανεξάρτητη διερεύνηση για εξοδικαστικές εκτελέσεις και οι παραβάτες πρέπει να αρθούν να ενώπιον της δικαιοσύνης. Πρέπει να καταδικάσουμε επίσης την επίθεση στο Τζαβαχά και να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους των θυμάτων. Τέλος, είναι σημαντική και μεγάλη η ανησυχία μας για τις διώξεις που υφίστανται ορισμένες θρησκευτικέ ομάδες στο Ιράν. Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μπορεί να γίνει μονάχα εφόσον ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα των ομάδων αυτών και των περιοχών αυτών. Ευχαριστώ κύριε Ρομπέ Βαϊρουέδα. Τώρα οι εκπρόσωποι των ε, πολιτικών ομάδων. Πρώτος ο κύριος Σόνικ του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχει λεχθεί και σε προηγούμενη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2010 κρίθηκε ένοχη συνωμοσία η Νασρίν Σότουντε στο κράτος του Ιράν και συνελήφθη για τέσσερις μήνες. Τώρα καταδικάστηκε σε ενδεκαετή κάθερξη καθώς επίσης στερήθηκε την άδεια άσκηση επαγγέλματο για 20 χρόνια και επίσης δεν μπορεί να αποχωρήσει από το Ιράν. Και άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι, σε άλλους πολιτικούς κρατούμενους επευλήθησαν βαριές ποινές κάθερξης. Πρέπει να αντιταχθούμε σε τέτοια παραδείγματα παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων. η Νασρίν Σοτουντέ έχει αφιερώσει την ζωή της στην υπεράσπιση ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο επειδή συμμετείχαν σε δημοκρατικές ε, ομάδες. Δεν μπορούμε να μείνουμε άπρακτοι όταν βλέπουμε αυτά τα τεκτενόμενα εκεί. Κρέτου, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ. Το να ζητούμε την άμεση απελευθέρωση της Νασρίν Σαρουντέ και όλων των πολιτικών κρατουμένων στο Ιράν είναι νομίζω κάτι που οφείλουμε. Χιλιάδες Ιρανοί πλήρωσαν με τη ζωή τους το ότι εξέφρασαν την διαφωνία τους σε σχέση με το καθεστώς που κυβερνά. Καταδικάστηκε σε 11 ε, χρόνια κάθερξης η Νασίνη Σοτουντέ μετά από την ε, πολύμηνη απομονώση της στη φυλακή επειδή υπερασπίστηκε ανθρώπους που είχαν διαφωνήσει με την ε, κυβέρνηση. Και όπως πολλοί αντιφρονούντες στο Ιράν υποφέρει υποφέρει μαζί με όσους εξέφρασαν την άποψή τους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποδείξει την αλληλεγγύη της και την δέσμευσή της να, πάυσει, να, να ζητήσει να πάψουν τέτοιες δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να δείξει την αποφασιστικότητά της ώστε όλες αυτές οι παραβιάσεις να πάψουν. Ο κύριο Τάνοκ από του Ευρωπαίου Συντηρητικού και Μεταρρυθμιστέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ στο ζώμα αυτό ότι η ελευθερία έκφραση και διαφωνία που εμεί απολαμβάνουμε ω δεδομένο δικαίωμα στην Ευρώπη κάπου λείπει ή δεν υπάρχει και καθόλου σε άλλα μέρη του κόσμου. Σήμερα συζητάμε το Ιράν. Για άλλη μια φορά ε, μιλούμε για το πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση σε μια Ισλαμιστική δημοκρατία. Ω δικηγόρο, η κυρία Σοτουντέ ε, ενίσχυσε πολλού από του αντιφρονούντε ε, που κατηγορήθηκαν μετά τι εκλογέ και τα βία επεισόδια πριν από 18 μήνε. Ήταν ερωικό το έργο τη σε μια χώρα που εκτελεί στιγνά ακόμη και παιδιά. Εδώ λοιπόν η εξαπλωνόμενη προπαγάνδα για απειλέ κατά τη ασφάλεια του κράτου είναι κάτι που το καταπολέμησε ε, με 11 χρόνια κάθριξη δεν μπορεί πλέον να ασκήσει καν το επάγγελμά τη ω δικηγόρο. Θα πρέπει να απελευθερωθεί χωρί όρου και θέλω, είπατε εκπρόσωπο, να προβάλλει αυτό το αίτημα. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου μιλά για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τι βίαιε ενέργειε του καθεστώτο του Αχμαντινετζάτ. Θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε τη χώρα αυτή όχι μόνο από την άποψη των εμπορικών μα συμφερόντων αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκο, κύριο Σκουρίο. Σκουρία για ένα λεπτό. Stiamo affrontando, signor Commissario, l'ennesimo dibattito. Εμείς από τις πολλαπλές μας ε, για την παραβίαση της δημοκρατία στο Ιράν. Πρόκειται αυτή τη φορά για μια δικηγορίνα που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν. Έτσι χτυπάτε, χτυπιέται το πρόβλημα στη ρίζα του. Δηλαδή δεν ε, χτυπάμε κατευθείαν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε λίγες εβδομάδες πάλι θα είμαστε εδώ μέσα για να μιλάμε για μια ακόμη περίπτωση ενό στοιχειώδους ανθρωπίνου δικαιώματος στο Ιράν. Θα μιλάμε για δραστηριότητα κατά της ασφάλειας, προπαγάνδα κατά του καθεστώτος και οποιοδήποτε άλλο φτιαχτό έγκλημα. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κόψει εντελώς τις σχέσεις της με αυτό το καθεστώς το οποίο παραβιάζει όλες τις αρχές που βασίζονται που βασίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος Κάρη. Για άλλη μια φορά, μια αποκρουστική κατάσταση συμβαίνει στο Ιράν. Μιλήσαμε πριν από τα Χριστούγεννα για, τον, για την Άστιανη η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο διαλυθοβολισμού η δίθ δίθεν για αμυχία και συμμετοχή σε φόνο. Σήμερα έχουμε παρόμοια υπόθεση της Νασρίν Σότουντέ που καταδικάστηκε σε 11 χρόνια κάθριξη επειδή έκανε τη δουλειά της. Της πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία. Ο σύζυγός της συνελήφθη ακόμα μέσα σε αυτή την εβδομάδα για διασπορά ψευδών. Άντε τώρα βγάλε άκρη. Πρέπει να ασκήσουμε κάθε δυνατή επιρροή που διαθέτουμε για να σταματήσει αυτή η παραφροσύνη και αυτή η βαριά κακομεταχείριση ιδίω των γυναικών. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κέλλη, ο Κούτας. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η καταδίκη της μεταχείρισης στη Μάλλον η καταδίκη της ε, κυρίας Τουντέ δείχνει πόσο δεν υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο Ιράν. Από το 2009 με την εκλογή του κυρίου Αχμαντινετζά τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται ακόμη πιο κατάφορα και πολλοί είναι εκείνοι που καταδικάστηκαν, διώχθηκαν γιατί διαφωνούν με το καθεστώς. Η, ε, κάθριξη, φυλάκιση 11 ετών, η ποινή για 11 ετή κάθριξη της κυρίας Σοτουντέ οφείλονται όχι μόνο στη διαφωνία τη με τα αποτελέσματα των εθευμένων εκλογών του 2009, αλλά γιατί υπερασπίστηκε και ανθρώπου που ήδη είχαν διωχθεί από το καθεστώ. Αυτό δείχνει πόσο δεν μπορούν οι δικηγόροι να κάνουν χωρί παρεμβολέ τη δουλειά του στο Ιράν. Και είναι και μία σαφή ε, περίπτωση όπου βλέπουμε ότι κανένα κράτο δικαίου δεν εφαρμόζεται. Κύριε, ε, θέλουμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή κανένα είδο συνεργασία οικονομικών να μην υπάρχει με το Ιράν μέσα από αυτέ τι συνθήκε. Ευχαριστούμε ο κύριο Τσαρνέτσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πρόεδρε, εδώ έχουμε άλλη μια περίπτωση που πραγματικά σκανδαλίζει την ε, ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και εμάς τους βουλευτές. Εάν εφαρμοστούν ε, οι ποινές όπως έχουν αποφασιστεί ε, το Ιράν θα είναι το μόνο κράτος για το οποίο δεχόμαστε να συνεχίζουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα ισχύει πλέον καμία από τι γνωστέ δημοκρατικέ αρχέ, καμία από τι διεθνεί προδιαγραφέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε λοιπόν από τη μια να έχουμε εμπορικέ σχέσει και από την άλλη ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, Ορθώ το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζει το ζήτημα αυτό. Πρέπει να ασκηθεί πολιτική πίεση. Έχουμε άλλη μια περίπτωση όπου με τη δράση μας στο τώρα Ευρωκοινοβούλιο δεν έχουμε υπάρξει αποτελεσματική στο να πιέσουμε το Ιράν. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όσοι αγωνίζονται υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ιράν υφίστανται διώξεις από πολλά χρόνια η υπόθεση της κυρίας Σοτουντέ εντάσσεται σε αυτές τις διώξεις. Στρέφεται το Ιρανικό καθεστώς κατά των λίγων εκείνων δικηγόρων οι οποίοι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίδιες συνέπειες θα υποστούν και άλλοι. Οι δικές μας προσπάθειες να επηρεάσουμε την κατάσταση δεν καρποφορούν. Νομίζω ότι η κυβέρνηση που ασκεί την εξουσία στη χώρα αυτή είναι απολύτως αυταρχική και ο μόνος τρόπος είναι να ασκήσουμε πολύ εντονότερη πίεση στην Ιρανική κυβέρνηση για να επιτρέψει στους Ιρανούς να αναπνεύσουν πιο ελεύθερα. Εσάγια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Νασίν Σοτουντέ είναι από τους πλέον γνωστούς συνηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Έχει υπερασπιστεί και ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά στα δικαστήρια, ακόμα και ανήλικοι, οι οποίοι δεν είχαν διαπράξει κανένα δίκημα. Πρόκειται για ένα βάρβαρο καθεστώς ταραχές που σημειώθηκαν προ στο Ιράν οδήγησαν τις Ιρανικές αρχές να επιβάλλουν πολύ βαρύτερα μέτρα κατά των ε, ακτιβιστών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει και σχετικές δηλώσεις. κυρία Ντε Όντενμπεργκ. Σας ευχαριστώ. Στη διάρκεια της προηγούμενης συζήτησης για θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν πριν από λίγους μήνες, σας είχα δηλώσει τότε ότι καθημερινά πέντε πολίτες του Ιράν πληροφορούνται ότι πρόκειται να χάσουν τη ζωή τους σύντομα στην βάση θανατικών καταδικών που εκδίδουν τα δικαστήρια. Η Νασέν Σοτουντέ συνελήφθη στις 4 Σεπτεμβρίου, βασανίστηκε, καταδικάστηκε και είναι ξεκάθαρα ένα παράδειγμα τέτοιων υποθέσεων που σας θυμίζω τον Μοχάμεντ Ισίμ Ισλαντέχ που έχει καταδικαστεί σε 9 χρόνια κάθριξη. Άλλος δικηγόρος πρόκειται να περάσει ένα χρόνο στη φυλακή μόνο επειδή υπερασπίστηκε τον πελάτη του ενώπιον του δικαστηρίου. Νομίζω ότι πρέπει να ζητήσουμε από την ύπατη εκπρόσωπο να επιμείνει και να περιλάβει τα θέματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων ε, στο διάλογο με το Ιράν. Μακοβέη. Η Νασρίν στο Τουντέ είναι μια πολύ σοβαρή δικηγόρος και μια πολύ σοβαρή περίπτωση. 11 χρόνια κάθεξη ε, απαγόρευση να ασκήσει το επάγγελμά της και ε, πάγωμα των περιουσιακών της στοιχείων. Τι έκανε. Ε, υπερασπίστηκε την κυρία Αχμαμπάντη και άλλους που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για λόγους ε, ε, διαφωνίες με το καθεστώ. καθεστώς. Το 2009, 15 δικηγόροι που έχουν περασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταδικαστεί και έχουν φυλακιστεί στο Ιράν. Αυτά είναι μέτρα που παραβιάζουν κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου. Ζητώ από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρέμβουν και να πετήσουν την άμεση απελευθέρωση της Νασρίνης Ατουντέ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο Επίτροπος Φίλε. Αν μπορείτε να απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα και να κάνετε την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί ιδιαιτέρως για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Τα προηγούμενα δύο χρόνια η συνθήκες από το κακό πήγαν στο χειρότερο. Είναι πλέον ανυπόφορε για όσου εργάζονται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Η Νασρίν Σοτουντέ και άλλοι πολλοί όπω εκείνοι που ε, αγωνίζονται για να υπερασπιστούν τα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Είναι σαφές ότι όσοι στο Ιράν είναι αρκετά ε, γενναίοι ώστε να υψώσουν το ανάστημά τους κατά των καταπιεστών τους, ε, διακινδυνεύουν να πέσουν θύματα εκφοβισμού, να φυλακιστούν ή και χειρότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υψώνει τη φωνή της. Δέκα δηλώσεις ε, δημοσιεύτηκαν το 2010 τις ε, εξέφρασε και τις παρουσίασε η ύπατη εκπρόσωπος η κυρία Άστον για παρόμοιες περιπτώσεις αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίστηκε και σε άλλες περιπτώσεις ανθρώπους στο Ιράν οι Ιρανικές αρχές κλήθηκαν να δώσουν στοιχεία, να αποσαφενήσουν κάποιες περιπτώσεις και να βελτιώσουν την κατάσταση στη χώρα. Η υπόθεση της Ρασίντο Τουντέφ σήμερα για την αντιπρόεδρο την κυρία Άστον ε, έχει γίνει από τις 14 Ιανουαρίου 2011 αντικείμενο δήλωσης. Λέει ότι και εκείνη και η κυρία Ζαράη που είναι δημοσιογράφος και δημοσιογράφος και έχουν καταδικαστεί και σε... η μία σε 11 και άλλη σε 4 χρόνια κάθριξης δεν είναι κάτι που μπορεί να είναι αποδεκτό. Μιλάμε για το μέλος του Ιράν που εξελέγει σε επιτροπή του ΟΗΕ για να εκπροσωπεί τη χώρα της. Ε, μιλάμε για δύο ανθρώπους που τους έχουν ε, αφαιρεθεί τα βασικά τους δικαιώματα, βασικέ τους ελευθερίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να θυμίζει στις Ιρανικές αρχές ότι πρώτο τα απ' όλα, πρωτίστως, πρέπει να συμμορφώνονται με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις ε, συμβάσεις και τις συμφωνίες, τις οποίες οι ίδιοι υπέγραψαν και κύρωσαν θα πρέπει να αναζητούμε τρόπους ώστε η δράση μας και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν να γίνουν αποτελεσματικότερες, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο λαός του Ιράν αξίζει ε, το καλύτερο. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Επίτροπε, η συζήτηση λίγη. Διαδικαστικό. Πολύ σύντομα. Στο Κοινοβούλιο. Έχουμε μία εντελώς επιφανειακή ομάδα εργασίας για το πώς θα αναδιοργανώσουμε τις εργασίες της Ολομέλειας. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο την Πέμπτη το απόγευμα και αυστηρούς προέδρους, όχι τόσο αυτάρεσκους, για να μπορούμε να έχουμε πιο ενδιαφέρουσες Ολομέλειες. Να το πείτε στον κύριο Σβόμποντα, κύριε Πόσελτ, που προεδρεύει στην ομάδα εργασίας Ψηφίζουμε. Πάρτε τις κάρτες ψηφοφορία σας, παρακαλώ. Έχω 7 προτάσεις για ψηφίσματα για το Πακιστάν. Θα ψηφίσουμε πρώτα για το Πακιστάν.